τροπολογία. Εγώ λοιπόν πρέπει να την απορρίψω. Και νομίζω ότι πρέπει να την απορρίψουμε όλοι. Okay. Μάλιστα. Ποιοι λοιπόν διαφωνείτε, αν μπορείτε να σταθείτε όρθιοι για να δούμε πόσοι διαφωνούν. I think it's more than, more than enough. Νομίζω ότι είναι περισσότεροι από 10, είστε περισσότεροι από αρκετοί. Ψηφίζουμε λοιπόν για το ψήφισμα υπέρ, κατά, Αποχές. Η τροπολογία έχει απορριφθεί, εξ όσων κατάλαβα. Αποσύρθηκε διότι περισσότεροι από 10, περισσότερα από 10 μέλη που βρίσκονται παρόντα στην Ολομέλεια την ε, απέρριψαν. Ψηφίζουμε λοιπόν για το ψήφισμα στο σύνολό του. Κοινή πρόταση ψηφίσματο συνολικά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το επόμενο σημείο που θα ψηφίσουμε είναι το θέμα του Αζερμπαϊτζάν. Και πάλι ψηφίζουμε τις έξι προτάσεις ψηφίσματος. Πρώτα απ' όλα, το ψήφισμα της ΓΚΟΕ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την κοινή πρόταση ψηφίσματος. Συνολικά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέλος, ψηφίζουμε για τη Λευκορωσία. Και πάλι έξι προτάσεις ψηφίσματος για την Λευκορωσία. Προηγουμένως όμως έχουμε πρόταση ψηφίσματος και πάλι ξεχωριστή της ΓΚΟΕ. Υπέρ της πρότασης του, του ψηφίσματος της ΓΚΟΕ. Κατά αποχές προφανώς απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την κοινή πρόταση τώρα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. να ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Προφανώς και εγκρίνεται. Οπότε συνάδελφοι, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος για την προσέλευσή σας και την παρουσία σας. Ως προς τις ανακοινώσεις, από την ομάδα των φιλελευθέρων ζήτησα κάποιες είχα κάποιες αιτήσει διορισμού στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και αντιπροσωπείες και αυτές οι αιτήσει θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Αν δεν υπάρξουν διορθωτικές παρατηρήσεις μέχρι την υποβολή των πρακτικών, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά. Τέλος, να να κηρύξω τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης. μάλλον για τα ψηφίσματα της σημερινής ε, συνόδου θα γνωστοποιηθούν αμέσως τις ενδιαφερόμενες άρχες λήξη της συνεδρίασης καλό ταξίδι στις χώρες σας.